βούλευση για το μέλλον της πόλης και ότι οι απόψεις θα ληφθούν υπόψη από τις αρχές. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον Επίτροπο Χάν. Κατόπιν αυτού υπάρχουν έξι ψηφίσματα τα οποία έχουν υποβληθεί. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση και αρχίζει η ψηφοφορία. Καταρχήν για το Πακιστάν ή τουλάχιστον το κοινό ψήφισμα των έξι πολιτικών ομάδων χωρίς τροπολογίες. Παρακαλώ να ψηφίσετε. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές το ψήφισμα έγινε αποδεκτό. Ερχόμαστε τώρα στη Λευκορωσία και εδώ υπάρχει ε, κοινό ψήφισμα. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, και αυτό το ψήφισμα εάν ε, βλέπω καλά έγινε ομόφωνα αποδεκτό σύμφωνα με ε, την ημερήσια διάταξη έχουμε τώρα την κατάσταση πολιτιστική κληρονομιά του Κασκάρ με μία τροπολογία ποιος είναι υπέρ αυτής της, ε, αυτού του ψηφίσματος κατά απορρίπτεται η αίτηση τροπολογίες και τώρα γίνεται ονομαστική ψηφοφορία για την υιοθέτηση του κοινού ψηφίσματος. Συμμετείχαν όλοι. Τότε κλείνουμε. με 26 ψήφους υπέρ, μία κατά και πέντε αποχές ε, έγινε αποδεκτό το ψήφισμα. Από το Συμβούλιο έλαβα την ε, θέση του Συμβουλίου και την θέση Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τώρα ε, έχει τρεις μήνες το Κοινοβούλιο χρόνο να αποφανθεί μέχρι τους επόμενους τρεις μήνες και ε, τα πρακτικά θα υποβληθούν ε, προς ε, αποδοχή.